Ε, ευχαριστούμε και ξεκινάμε συνεδρίες. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ράιμακ που μας εγκαταλείπει για να αναλάβει νέα σημαντικά καθήκοντα. Ε, θα αναλάβει τη θέση του πρέσβη της ε, Δημοκρατίας της Τσεχίας στην Μόσχα. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ναι, τα είπατε ήδη. Ε, ορίστηκα πρέσβης της Τσεχίας στην Μόσχα και χθες υπέγραψα τα σχετικά έγγραφα ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Κοινοβουλίου, άρα στις 16 Δεκεμβρίου, 16 Δεκεμβρίου, Δευτέρα, θα πάψω πια να είμαι συνάδελφό σας. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία θα πρέπει να ολοκληρώσουμε πριν το τέλος της θητείας. Ήταν εξαιρετικά πολύτιμη η εμπειρία μου εδώ, ήταν μια ανθρώπινη εμπειρία και όλα αυτά θα τα μεταφέρω μαζί μου στη Μόσχα. Εύχομαι σε όλους κάθε επιτυχία, καλή επιτυχία και για τις ε, μελλοντικέ ευρωεκλογέ. και αν τύχει να βρεθείτε στη Μόσχα, μην ξεχνάτε πως ένας από τους συναδέλφους σας θα είναι εκεί και είστε πάντοτε ευπρόσδεκτοι να έρθετε για καφέ. να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς μας ε, γιατί χάρη σε εκείνους ήμουν ε, ε, μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Un caro saluto. Θερμούς χαιρετισμού λοιπόν από όλη την Επιτροπή στο συνάδελφο Ρέμεκ. Δεν αποκλείεται κάποιος από εμά να δεχτεί την πρόσκλησή σας. Σας ευχόμαστε καλή δουλειά, καλή επιτυχία και Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας ε, στην Επιτροπή. Ε, όπως ξέρετε, τις προάλλες είχαμε και τον διορισμό της συναδέλφου Κολάρισκα Μπομπίσκα στο Υπουργείο Έρευνας της Πολωνίας. Οπότε, εδώ στα τέλη της θητείας η Επιτροπή μας αλλάζει σημαντικά. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Ψηφίζουμε λοιπόν, κάνουμε μια δοκιμή. Για δοκιμάστε όλοι να δούμε αν δουλεύουν όλε οι κάρτε. Avete ε, Ψηφίσατε όλοι. Εντάξει, δουλεύουν τα μηχανήματα. τέλο τη ε, ψηφοφορία. Είναι όλοι παρόντε, όλα εντάξει. Ωραία. Non funziona. Δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Λοιπόν, αλλά ξέχασα την κάρτα μου. Πρόεδρε, πρόεδρε. Αν κάνουμε άλλη μια δοκιμή. Ψηφίστε παρακαλώ. Ωραία, τέλο ψηφοφορία. Μεσή Ο κύριο Μπουτικόφερ. Το μηχάνημά μου δεν λειτουργεί. και Λοιπόν, για ε, δοκιμάστε άλλη μια φορά. Η macchina funziona. Όχι. Δεν λειτουργεί, το μηχάνημα τώρα. It's okay? Encore un test. Ακόμα μια δοκιμή. Άλλη μια δοκιμή λοιπόν. Ας ψηφίσουμε άλλη μια φορά. Εντάξει τώρα, λειτουργούν όλα. Τέλεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. Ραπόρτο Βαλεάν. Αφαβόρε. Έκθεση Βαλεάν. Υπέρ της συμβαστικής κατά αποχές εγκρίνεται. Έκθεση του Ζενόφσκι. Υπέρ τη συμβαστική κατά αποχές εγκρίνεται. Έρτζοκ. Έκθεση Χέρτζοκ. Ας ξεκινήσουμε. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Από κοινού 25, 26, 27, 28 και 29. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνονται. 66. Υπέρ. Κατά. Ας κάνουμε μια δοκιμή. Είναι διαφορετική αίθουσα, είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την 66 τη συναδέλφου Τικάου. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 26 κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 76 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 77 και 78 μαζί υπέρ κατά <clears throat> αποχές νομίζω πως εγκρίνεται. Ας κάνουμε μια επαλήθευση τροπολογίες 77 και 78. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 79 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ.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 87 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111. 111. Είναι σωστό. Εγκρίναμε την 109, γι' αυτό περνάμε στην 111, εντάξει. Όλοι συμφωνείτε, ωραία. 111 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15, ε, τροπολογία 127 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 130 υπέρ κατά Έλεγχος για την 130. Ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 18 κατά, εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές. Έλεγχος. Ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτή η αίθουσα δεν με δεν μπορώ να μετρήσω υπέρ. Κατά... Α, ναι, ηλεκτρονική ψηφοφορία κάνουμε, συγγνώμη. Τέλος ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 140. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100, ε, συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές... Α, κάτι ξέχασα. Συγγνώμη. Ε, είναι η 150. Τροπολογία 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 155 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Τέλος. Τήρεται υπέρ. Εγκρίνεται. 160 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ. όχι, όχι. Και την 100, και 162 έχει καταπέσει. Ωραία. 163. 163 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχέ ε, εγκρίνεται. τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, μου 40, 40 όχι 47, η 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά για όλες τις τροπολογίες που εγκρίναμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. 47 υπέρ, 4 κατά, μία αποχή. Και τώρα για το νομοθετικό ψήφισμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται για τις διαπραγματεύσει. Ψηφίζουμε πάλι. Ωραία. Τέλος της ψηφοφορίας. 39 υπέρ, 8 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στη συνάδελφο. Και περνάμε στην έκθεση Μπουτικόφερ. Παρακαλώ. Για τον, για τη συμβαστική πρόταση 56. Δεν θέλω να βάλω το όνομά μου για αυτή τη συμβαστική πρόταση. Τίτλο 1. Ξεκινάμε λοιπόν. Τίτλο 1. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση ηλεκτρονική. Παρακαλώ, ψηφίστε. τίτλος 1, OD, ψηφίζουμε τέλος της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, 5, 6 μαζί, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 και 14 μαζί. Υπέρ. Κατά <clears throat> αποχές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 κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε επαληθεύουμε για 23 Τέλος ψηφοφορίας 31 προς 18. Εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήθελα να σας κάνω μια πρόταση, αν συμφωνείτε, να ψηφίσουμε από την 25 στις 40 unblock. Α, από την 25 μέχρι την 36. Όχι. Ποιος διαφωνεί. 25 με 35 συμφωνείτε. Όλοι. Όχι. Ε, εντάξει, τώρα τις ψηφίζουμε. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται.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 Τέλο ε, Κιούζα. Τέλος της ψηφοφορίας. 27 και 28 απορρίπτονται. 27 προς 28 απορρίπτονται. 37 ε, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 ρούμπι κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για την 52. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Τέλος της πληροφορίας. 29 προς 21 εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές κατά κατά ε, στο κατά είμαι. Απορρίπτεται. Για την 11 να ελέγξουμε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. 24 υπέρ 30 κατά απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 σε δύο κομμάτια το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κατά τη γνώμη μου αλλά θα κάνουμε μια, έναν έλεγχο για την 71 πρώτο τμήμα τέλος της ε, ψηφοφορίας 30 υπέρ άρα εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται ας κάνουμε άλλη, άλλο ένα έλεγχο για το δεύτερο κομμάτι της 97 η, τέλος της ψηφοφορίας 31 προς 22 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 165 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22 παρακαλώ Τέλος της ψηφοφορίας, 38 προς 16 εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14. Α, όχι. Υπάρχουν δύο τέσσερα. Ωραία. 4 της Ρέτζη. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ. Τα αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 199 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 202. Α, 19. 19 συμβιβαστική έλεγχος. Οι δικοί μου καταψηφίζουν. Τέλος της ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. 202 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 ένβη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 242 ε, υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 244. Α, θέλετε έλεγχο για τη 242, παρακαλώ. Τέλος της πληροφορίας. 25 υπέρ, 28 κατά. Απορρίπτεται. 244 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 246 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 258 και 257, όχι, 58, 258 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για τη 258. Κιούζα. Τέλος ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 21 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ κα... Παρακαλώ, κύριε Μπουτικόφερ. Πρόεδρε, ψηφίσαμε το 257. Α, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Συγγνώμη, εντάξει, κατάλαβα. Ωραία. Την 26 τη συμβαστική την ψηφίσαμε. Πάμε στην συμβαστική 27. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 271 δεύτερο τμήμα υπέρ από τη 271 ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 275 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 276 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 29 υπέρ κατά ναι 29 29 όχι 9 που είπα 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 281 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 283 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 284 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται κατά τη γνώμη μου, αλλά στο ελέγξουμε. Για τη 284, παρακαλώ, ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 34-17. 286 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 287 πρώτο τμήμα υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 287 δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 288 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 289 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 295 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 ε, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 302 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 303 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 304 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 300 Α, ίσως να απορρίπτεται. 304 να ελέγξουμε. 304 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ε. Τέλος ψηφοφορίας. 20 προς 34. Απορρίπτεται. 306. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. 307. 5 τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πέμπτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 32 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 με προφορική προσθήκη ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 324 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 330 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 331 σε δύο τμήματα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 332 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 333 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 334 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 335 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 34, 35 και 36. Ποιος είναι υπέρ, μαζί. Κατά, αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 35, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 340 σε δύο τμήματα, υπέρ. Πρώτο τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 341 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 342 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 343 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 344 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 345 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 38. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 352 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 353 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 355 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 358 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 359 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 364 υπέρ, σε δύο τμήματα, συγγνώμη, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 43. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 62. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 369. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 370. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 371. Υπέρ. Κατά αποχές Ηλεκτρονικό έλεγχο παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Δίνουμε μια ευκαιρία στην κυρία Τόια. Τέλος ψηφοφορίας. 20 προς 32. Απορρίπτεται. 3.72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 374 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 377 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 378 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 379 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα, τροπολογία 1 της Επιτροπής Απασχόλησης, δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 384 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 385 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 387 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 392 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 399 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 402 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 407 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σε δύο τμήματα, συγγνώμη, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Συμβαστική τροπολογία 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεστική τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 424 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 429 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 430 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 54 υπέρ. Α, συγγνώμη, διορθώνει ο Πρόεδρος. Η τροπολογία 20 της Επιτροπής Περιβάλλοντος καταπίπτει, δεν ψηφίζουμε. Συμβαστική τροπολογία 54, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 452 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 453 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 56. Η άλλη απέσυρε την υπογραφή της υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για τη συμβαστική τροπολογία 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Τέλος υπήρχε μία ψήφος ε, που περίσευε. 41 ψήφοι υπέρ, 8 κατά, εγκρίνεται. Η συμβαστική τροπολογία 56. Τροπολογία, ε, συμβαστική 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 486 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 494 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 495 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 496 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 497 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 498 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 499 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 500 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 506 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 507 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 509 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά η ψηφοφορία Votazione chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. 45 υπέρ, 5 κατά και 5 αποχές. Εγκρίνεται, συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Και περνάμε στην επόμενη έκθεση. La collega... Τη συναδέλφου Βαλεάν. Τροπολογία 12. <coughs> υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τελική ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλο ναι. le ναι. Τέλος ψηφοφορίας. 50 υπέρ, 1 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Emendamento 4 e 5. Τροπολογίες 4 και 5 από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική 4, συμβαστική 5. Contrari, astenuti, appro... Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται unblock 7, 8, 9 και 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται Α, να το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ 7, 8, 9 και 3 του budget ε, τέλος της ψηφοφορίας 34 υπέρ, 18 κατά εγκρίνεται 31. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 6. Συμβαστική 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογίες 37 και 38 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Ε, τροπολογία 73. Όχι. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Budget 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε, τροπολογία, συγγνώμη, 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 45 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ε, προϋπολογισμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70... 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 όχι, 70, 70 έχει καταπέσει. Δεν την ψηφίσαμε. Περάσαμε από το 71 στο 72. 74 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. 49 υπέρ, 1 κατά. Εγκρίνεται. για την νομοθετικό, νομοθετική πρόταση ε, υπέρ και μάλλον ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τέλος 50 υπέρ ένας κατά και τώρα για τη διαπραγμάτευση ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ τέλος της ψηφοφορίας 49 υπέρ, δύο αποχές, μάλλον δύο κατά μία αποχή, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Και τώρα περνάμε στην ε, εισηγήτρια Ουλσκοκ. Παρακαλώ λίγο ακόμα προσοχή για να τελειώσουμε. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβεβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε μια επαναλήθευση για την 51 Τέλος ψηφοφορίας. «31 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Tutti. Ma io devo togliere questo. Cosa? credevo visto qualche voto di dissenso che cambiavano le cambiavano. Chiuso, chiuso. 51 a favore, uno contrario. 51 υπέρ, 1 κατά, κανένα, καμία αποχή, συγχαρητήρια. Έκθεση Μπέντστεν. 35 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 40 υπέρ. Συμβαστική 3 μάλλον για έλεγχο. Ψηφίζουμε. Chiusa. 35 a favore, 17 contro. 35 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. 40, τροπολογία 40. Contrari, αφαιρούνται respinto. Ε, αποχές εγκρίνει, απορρίπτεται 41 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά, αποχές ε, απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίν, ναι, απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές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 κατά αποχές εγκρίνεται 61 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απόρριπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 έλεγχος ηλεκτρονικός για την 72 παρακαλώ Χιούζα Πέρας ψηφοφορίας 18 υπέρ 29 κατά απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές Α, συγγνώμη, αφαιρέθηκα. 73, 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 76 το δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 και 84 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ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 Αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά. Αποχές απο... Ε, εγκρίνεται υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 25 ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τελική ψηφοφορία. Οτοκιούζα. Τέλος της ψηφοφορίας. 34 favore, 34 υπέρ 15 κατά, 2 αποχές και εγκρίνεται. Passiamo all'ultima votazione Τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. L'ultima votazione della mattinata. Un attimo ancora di attenzione e poi abbiamo finito. Τελευταία ψηφοφορία λοιπόν και α, τελειώσαμε. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Την 5 ξέχασα. Την 5 υπέρ, κατά, απόχέ, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, απόχέ. απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, απόχέ. Έλεγχο ηλεκτρονικό. Ψηφίστε παρακαλώ. Aperta. Non è aperta. Τώρα ψηφίστε, τώρα άρχισε η ψηφοφορία. Κιούζα. Τέλος της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3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 αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 4, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 35, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 36, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 5, με την προσθήκη το ΙΣΕΡ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται, τροπολογία 50, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Δεύτερο τμήμα Τη 67. Τέλος ψηφοφορίας. 36 υπέρ. 15 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 έχει απορριφθεί αλλά ας ελέγξουμε Έντεκα υπέρ 35 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Ευχαριστώ. 74 ε, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα 74, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Μάλιστα. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ε, της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα τώρα. απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 79 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται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 αποχές ε, απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λοιπόν ψηφίζουμε για την τελική ψηφοφορία votazione chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. 38 υπέρ, 7 κατά, ένα, μια αποχή, συγχαρητήρια. Τελειώσαμε και με τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και σήμερα ήμασταν αρκετά γρήγοροι. Καλημέρα σε όσους φύγουν. Πέντε λεπτά για να φύγουν όσοι είναι να φύγουν γρήγορα γρήγορα.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 se volete lasciamo 5 minuti dai riprendiamo i nostri lavori se i colleghi vogliono gentilmente Παρακαλώ, οι συνάδελφοι θα μείνουν να καθίσουν για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Grazie. Θα δώσω το λόγο στην Μαρίτα Ουλτσκοκ <laughs> για να εξετάσουμε την έκθεση αυτή που αφορά την επαλήθευση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές και την τροποποίηση του σχετικού κανονισμού. Ήθελα να περιμένω να βγουν όλοι για να σου δώσω το λόγο, ώστε να είμαστε ήσυχοι. Παρακαλώ τους συναδέλφους. Η κυρία Ουλσκοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι η διεθνή συναυτιλία είναι, αποτελεί εξαίρεση. Από τις, εξαιρείται δηλαδή από τους στόχους για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανέλθει στο ζήτημα αυτό και έτσι η Κομισιόν υπέβαλε πρόταση κανονισμού για την παρακολούθηση και την κοινοποίηση ή την παρακολούθηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από την ναυτιλία. Είναι πολύ θετική η την παρακολουθηση των εκπομπων διοξειδιου του ανθρακα απο αυτή και τα μέτρα που προτείνονται είναι απολύτως απαραίτητα ακριβώς για να καθοριστούν και οι στόχοι για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την ναυτιλία. Διακόπτη πρόεδρος και ζητά να κάνουν όλη ησυχία. Το ζήτημα είναι λοιπόν να λάβουμε μέτρα για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και το στόχος είναι να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι. Αν ωστόσο δεν υπάρξει διεθνή συμφωνία για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε διεθνές επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να υποβάλει πρόταση νομοθετήματο για τι του διοξιδίου του άνθρωπου από την ναυτιλία έω το 2015 το αργότερο. Στην πρόταση προτείνεται ένα χρονοδιάγραμμα για τη θέση σε ισχύ αυτού του κανονισμού και όποιο δεν... εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικά ε, μεγάλη η προθεσμία αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να δράσουμε πιο γρήγορα. Ιδιαίτερα η Σύνοδος για το Κλίμα στη Βαρσοβία απέδειξε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πίσω από τους πολύ φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει προτείνει να εγκριθούν τα λευτικά σκάφη με όγκο μικρότερο από 5.000 τόνους. Εγώ διαφωνώ. Επίσης πιστεύω ότι ο κανονισμός θα πρέπει να επιβραβεύει εκείνες τις ε, μεθόδους που έχουν ήδη αξιοποιηθεί για την μείωση, τη δραστική μείωση των εκπομπών. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό τα σκάφη να πρέπει να πληρούν τέτοιου είδους κριτήρια, να μειώσουν δηλαδή τις εκπομπές τους. Και θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό ότι η Κομισιόν ε, προτείνει το είδος της μέτρησης να μπορεί να επιλεγεί από τα ίδια τα σκάφη. Τα σκάφη δηλαδή μπορούν να επιλέγουν ε, τον τρόπο μέτρησης των εκπομπών τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρίτα. Τώρα θα δώσω το λόγο στους Σκιώδης και πρώτος ο κύριος Τζόρνταν. Η κυρία Τζόρνταν, συγγνώμη. Συμφωνώ με την εισηγήτρια που λέει ότι ένα μέρος της ευθύνης για τη μείωση των εκπομπών θα πρέπει να αναλυφθεί και από τις, άλλες, ε, από τις μεταφορές, τις αεροπορικές και τις θαλάσσιες. Ιδιαίτερα αφού το μερίδιο των εκπομπών ε, στις θαλάσσιες μεταφορές, θα αυξηθεί. Όπως είπε και η εισηγήτρια, θα πρέπει να υπάρξει μια διεθνή συμφωνία και ιδιαίτερα σημαντική είναι σε αυτό το τομέα μια τομεακή συμφωνία. Στην αντιπροσωπεία, ήμουν στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην ε, Βαρσοβία, συναντηθήκαμε και με τους εκπροσώπους της ΙΚΑΟ για, την, ε, για τις αεροπορικές μεταφορές, αλλά στον τομέα αυτό η ΙΚΑΟ δεν έχει επιτύχει ε, σημαντικά αποτελέσματα. Εδώ και πολλά χρόνια ακούμε τις ίδιες και τις ίδιες υποσχέσεις. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι το έτος 2015 είναι πολύ σημαντικό, διότι τότε θα δούμε σε ποιο βαθμό θα είναι δυνατή η λήψη παγκόσμιων μέτρων, ποια μονομερή μέτρα θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί θα πρέπει να δούμε πόσο φιλόδοξοι θα πρέπει να είμαστε. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να πούμε σε κάθε περίπτωση σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε, αλλά δεν θα πρέπει να προστρέξουμε. Στο όνομα της ομάδας μου υποστηρίζω ένα αποτελεσματικό και απλό σύστημα που θα μας αποφέρει το σημαντικότερο επίτευγμα που θέλουμε να επιτύχουμε χωρίς να υπάρχουν μεγάλα διοικητικά εμπόδια. Είμαι της άποψης ότι οι στόχοι μας θα πρέπει να είναι σαφείς και όχι κατακαιρματισμένοι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε την έκθεση και με περισσότερες παραμέτρους σε αυτή την πρώτη φάση δεν θα επιτύχουμε τους ε, επιθυμητούς στόχους. Το να επεκτείνουμε το σύστημα αυτό και σε άλλα αέρια δεν νομίζω ότι θα προσέθετε κάτι στο, στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε. Κύριος Γιώχαν. Θέλω και εγώ να συμφωνήσω με την εισηγήτρια και να μιλήσω σου ειδικά. Συμφωνώ με τα κύρια σημεία της, της έκθεσης, ωστόσο θεωρώ και εγώ σημαντικό να μπορούμε πρακτικά να μειώσουμε τις διακουμπές διοξιδίου του άνθρακα από την ναυτιλία, διότι τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά και από διεθνή άποψη, ενώ τη διεθνή ναυτιλία και τα λιμάνια, που είναι τομείς που είναι πολύ, πολύ συχνά πυκνοκατοικημένοι. Και από αυτή την άποψη έχουν επιπτώσεις και η, η, έχει επιπτώσεις και σε αυτές τις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Οπότε χρειαζόμαστε στόχους και σε διεθνές επίπεδο και θα πρέπει να το συνδυάσουμε αυτό με το γεγονός ότι οι εκπομπές αυτές είναι τόσο υψηλές σε αυτές τις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Πιστεύω επίσης ότι θα έπρεπε να εισαχθεί ένα σύστημα στο πλαίσιο του IMO. Αλλά κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο, διότι η διεθνής ε, ναυτιλία έχει επιπτώσεις μεν στο κλίμα, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα η Ανατολική θάλασσα, η Βαλτική θάλασσα είναι μια ιδιαίτερα ρυπασμένη περιοχή. Κατάγαμε από αυτή την περιοχή και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσουν καν οι συζητήσεις. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε και πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το σύστημα αυτό, διότι το ερώτημα είναι και αυτό, πώς θα ε, μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη και πώς θα μπορέσει να γίνει αποδεκτό από τους εταίρους μας. Διότι θεωρώ ότι αν δημιουργήσουμε πρόσθετα διοικητικό άχθος, δεν θα έχουμε επιτύχει το, ε, το στόχο που θέλουμε. Γι' αυτό πρέπει να αναλάβουμε και πρακτική δράση, να αναλάβουμε πρακτικά μέτρα ακριβώς για την εφαρμοσιμότητα του συστήματος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο τομέας ε, της ναυτιλίας. Θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να συνδέεται με τον IMO, αλλά αν σκεφτούμε ποιες θα είναι ε, οι πρακτικές εφαρμογές του συστήματος, θα πρέπει να συζητήσουμε με τους ενδιαφερόμενους. Πρέπει να καθορίσουμε συγκεκριμένους στόχους, μεν, αλλά θα πρέπει επίσης να συζητήσουμε Πώ από την πλευρά της δικής μας Επιτροπής θα μπορέσουμε να φροντίσουμε για την καλύτερη δυνατή πρακτική εφαρμογή του συστήματος. Και νομίζω ότι θα ε, συζητήσουμε με την εισηγήτρια για το ζήτημα αυτό και στο, στο άμεσο μέλλον θα, υποφε, θα υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλε σκιώδει παρόντε. Ε, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση. Ο κύριο Οντί έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι ειδήμων για το θέμα αυτό. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε συνετοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως και να τα περιπλέκουμε όλα. Η ναυτιλία είναι ο κλάδος που εκπέμπει λιγότερα καυσαέρια και διοξείδιο του άνθρακα. Τώρα, να επιβάλλουμε τόσες πολλές υποχρεώσεις στις ναυτιλιακές εταιρείες, ήδη έχουμε ελάχιστα πια σκάφη με ευρωπαϊκή σημαία. Α είμαστε λοιπόν πολύ συνετοί και προσεκτικοί σε αυτή τη νομοθεσία που προτείνουμε. Και μάλιστα μετά από διαβουλεύση με ενδιαφερόμενου, ε, ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να περάσουμε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Α προσπαθήσουμε επιτέλου ε, να είμαστε στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό Εμεί οι κινητήροι μοχλοί για να απεμπλέξουμε τη συμφωνία αυτή, για να διευκολύνουμε τα πράγματα για την ναυτιλία, γιατί τα περιπλέξαμε για τι οδικέ και σιδηροδρομικέ μεταφορέ. Εγώ είμαι κατά τη της ενίσχυσης της γραφειοκρατίας. Αν και συμφωνώ με τους μακροπρόθεσμους στόχους, ότι δηλαδή θα πρέπει να περιορίσουμε τις ε, εκπομπές διεξουδίου του άνθρακα. Αλλά δεν ξέρω για την αυτιλία η επιτήρηση και η γραφειοκρατία είναι ο κατάλληλος τρόπος, γιατί πρόκειται για ένα, τρόπο μεταφο... ένα είδος μεταφοράς, ένα τρόπο μεταφοράς που εκπέμπει ελάχιστο διοξίδιο του άνθρακα. Ευχαριστώ κύριος Πρόντι. Grazie Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ επιμένω στην ε, ιδέα μου ότι θα έπρεπε να απλοποιηθεί η διαδικασία και να υπόκειται στην καταβολή δικαιωμάτων εκπομπών τη στιγμή που το καύσιμο ή κάθε στεροκαύσιμο ε, τοποθετείται στην αγορά και άρα στην πηγή να γίνεται μια τέτοια, μια τέτοια εισφορά που είναι και απλή και εύκολα εφαρμόσιμη και που ανταποκρίνεται στην ανάγκη να υπόκειται κάθε χρήση στερεών καυσίμων στην απόκτηση ε, δικαιωμάτων εκπομπών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε Και αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, παρακαλώ. Σα <laughs> Thank you very much. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλή σας μέρα. Καταρχήν θα ήθελα να πω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θερμά ευχαριστώ προς την εισηγήτρια. Γιατί ήταν πολύ ε, καλή και επικοδομητική η έκθεσή της, το σχέδιο έκθεσή της και θα συμβάλλει πιστεύω σημαντικά στη συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο. Πριν ε, περάσω στις λεπτομέρειες και σε αυτά που μας είπαν οι συγγήτρικες και οι συγγητές, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Παρόλο που η ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 3 με 4% των παγκόσμιων εκπομπών, στην Ευρώπη είναι 4% των εκπομπών διοξίδια του άνθρακα. Φαίνεται μικρό το ποσοστό, αλλά αν συγκρίνουμε τις εκπομπές ναυτιλίας με τις εκπομπές σημαντικών βιομηχανικών κλάδων, ε, μιλάμε για 180.000 τόνους διοξείδιο του άνθρακα του χρόνου. Ε, περισσότερο δηλαδή από ό,τι η τσιμεντοβιομηχανία, τα δηληστήρια ή η χημική βιομηχανία το χρόνο. Οπότε μην υποτιμάτε και την αυτιλία είναι σημαντικός τομέας εκπομπής διοξείδιο του άνθρακα και η ιδιαιτερότητά του οφείλεται σε αυτό που λέμε το low hanging fruits. Δηλαδή όλες οι μελέτες που γίνονται ε, και από εμά και από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό υποδεικνύουν ε, σημαντικό δυναμικό μείωση των εκπομπών μόνο με τη βελτίωση της ε, ενεργειακής απόδοσης των πλοίων και μάλιστα της τάξης του 25 με 75%. Τεράστιο δυναμικό οικονομίας δηλαδή και μείωση των εκπομπών και μάλιστα με σημαντική σχέση κόστους-οφέλους, δηλαδή οι επενδύσεις που θα γίνουν θα αντισταθμιστούν από σημαντικά κέρδη και ωφέλη. Και σε κανέναν άλλο τομέα, ούτε καν ε, στις οδικές μεταφορές ούτε στη βιομηχανία δεν μπορούμε με τόσο λίγο κόστος να έχουμε τόσο θεαματικά αποτελέσματα όσο στην αυτιλία σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική στρατηγική, όπως ε, περιγράφεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι μεσοπρόθεσμες φιλοδοξίες μας επιδιώκουν μέτρα μείωσης των εκπομπών που θα βασίζονται στην αγορά και που με επιτυχία έχουν εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς ή θα μπορούσε να, θα μπορούσε να βασίζονται σε προδιαγραφές αποτελεσματικότητας χρησιμοποιώντας αυτό το τεράστιο δυναμικό μείωση των εκπομπών χάρη στη βελτίωση τη ενεργειακή απόδοση των πλοίων. Και μάλιστα στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό στι αρχές του χρόνου ξεκίνησαν σχετικέ διαπραγματεύσει με πρόταση των Αμερικανών για μια σταδιακή προσέγγιση ε, σε ό,τι αφορά την εκπομπή αερίων από τα πλοία. Στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα ζήτημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές. Επίσης, δεύτερο βήμα θα είναι η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των πλοίων και η θέσπιση κάποιων στόχων αποτελεσματικότητας ως τρίτο βήμα, μακροπρόθεσμα ίσως και μέτρα που θα στηρίζονται στην αγορά. Όλες αυτές ε, οι προτάσεις έγιναν ευπρόσδεκτες από μερικές χώρες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όχι μόνο από χώρες της δύση. Η δύση ήταν αρκετά επιφυλακτικές, αλλά χώρες όπως η Σιγκαπούρη, ο Παναμάς, η Λιβυρία, αλλά και η Κίνα, που είναι χώρες με πολλά πλοία με δική του σημαία, είναι πρόθυμες να εξετάσουν κάποια μέτρα αποτελεσματικότητας, γιατί επαναλαμβάνω, οι επενδύσεις θα είναι πολύ αποδοτικές. Επενδύοντας στην απόδοση θα γίνουν πολύ μεγαλύτερες οικονομίες από ό,τι το ύψος των επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι για να ανταποκριθούμε στην εντολή που λάβαμε το 2008 στο πακέτο για το ενεργειακό και το περιβαλλοντικό κλάδο, οφείλουμε να προτείνουμε προτάσεις για να περιοριστούν οι εκπομπές ε, και της ναυτιλίας. Νομίζουμε ότι μια συνετή πρόταση μπορεί να ξεκινήσει με ε, παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακρίβωση. Έτσι θα δώσουμε περισσότερο περισσότερο χρόνο και στη διεθνή κοινότητα μέχρι το καταλήξει συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί η ναυτιλία είναι ο πιο ε, διεθνής κλάδος που υπάρχει. Και σίγουρα θα είναι πιο αποτελεσματικό τα προβλήματα να διευθετηθούν διεθνώς, αν γίνεται φυσικά. Η ΔΕΜΗ και αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες της συγκεκριμένης, ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε με σταυρωμένα χέρια για πάντα και κάποια στιγμή, αν υπάρξει παγκόσμια αδράνεια, ίσως θα μπορούσαμε να υποβάλουμε μέτρα μείωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο μεταξύ όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να αφήσουμε λίγο χρόνο στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για να εξετάσει όλα αυτά τα θέματα που ίσως καταλήξουν σε σημαντικά, και αποτελεσ... σημαντικά αποτελέσματα. Και ίσως το 2015 παρά είναι φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Τώρα, για τις άλλες προτάσεις που υποβλήθηκαν, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι μία από τις βασικές προ... προσεγγίσεις της πρότασης είναι μία προσέγγιση για ελάχιστη γραφειοκρατία και με την χρησιμοποίηση και αξιοποίηση υπαρχουσών τεχνικών και γράφων. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να ελέγξει τις εκπομπές εξετάζοντας ε, τα αρχεία που έχουν τα πλοία για την κατανάλωση καυσίμων και μάλιστα να τα κρατούν για πέντε χρόνια αυτά τα στοιχεία. Οπότε με την αξιοποίηση αυτών των στοιχείων θα έχουμε ελάχιστο κόστος ό,τι αφορά την υποβολή αυτών των στοιχείων και... για τα καυσαέρια. Τώρα αν δούμε πιο εξεζητημένε μεθόδους για την καταγραφή των εκπομπών, τότε χρειαζόμαστε συγκεκριμένο εξοπλισμό για την άμεση καταγραφή των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ή συγκεκριμένες ε, μετρήσεις ε, τη κατανάλωση καυσίμων για τα πλοία. Εκεί μπορεί να χρειαστούν και 50.000 ευρώ για τα ροόμετρα ή ίσω και πάνω από 100.000 ευρώ αν θέλουμε άμεση καταγραφή και καταμέτρηση των εκπομπών. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε τη βιομηχανία να εφαρμόσει τώρα τα πλούστερα και τα λιγότερα τα πανηρά μέσα. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. Η πρότασή μας περιορίζεται στους ε, μεγαλύτερους ε, εκπομπής, ε, δηλαδή σε πλοία κάτω των 5.000 τόνων ολικής χωρητικότητας και και καταναλώνται 40 με 45% του συνόλου των πλοίων. Νομίζω ότι είναι μια αναλογική λύση αυτή. Αλλά είναι και πολιτικό το θέμα. Ποια πλοία θα εξαιρεθούν. Θα μπορούσε κανείς να ζητήσει εναρμόνιση του πεδίου εφαρμογής με τις διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις. Και να καταλήξουμε στην απάντηση του 400 ίσως ήταν καλύτερη εναλλακτική. Για τα αλληλευτικά σκάφη θεωρούμε ότι δεν είναι πρόβλημα για τις εκπομπές διεξουδίου του άνθρακα και καλύπτουμε 25 πλοία ουσιαστικά από τα 10-11.000 πλοία που έχουμε τα αλληλευτικά. Και αυτά τα πλοία εκπέμπουν μόνο το 0,6% του συνόλου των εκπομπών διοξιδίου του στόλου. Μικρό ελάχιστο τμήμα δηλαδή. Και επιπλέον για τα αλληλευτικά σκάφη η εφαρμογή θα ήταν πολύ πιο επώδυνη σε σχέση με την ε, οδηγία που περιλαμβάνει μέτρα για τον έλεγχο από το σκάφος της σημαίας. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι κάλυψα τα περισσότερα σημεία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την ε, πλήρη ε, παρέμβαση και τώρα το λόγο έχει η συγγήτρια για να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω θερμά και την κυρία Γιόρδαν, και τον κύριο Πρόντι για τις επικοδομητικές τους προτάσεις. Νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Νομίζω ότι θα κάνουμε πρόοδο από κοινού. Τέλος, να πω ότι η διαδικασία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού είναι ο υπερκείμενος ε, οργανισμός και δεν μπορούμε βεβαίως να ε, ε, περιμένουμε όσο θέλουμε. Ίσως τελικά θα αποδειχθεί απαραίτητο να, αναλάβουμε, λάβουμε μέτρα από τώρα και νομίζω ότι αποδεικνύεται σαφώς πόσο δραματική είναι η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, ιδιαίτερα στα λιμάνια. Η Κομισιόν είπε ότι η βιομηχανία τσιμέντου και η χημική βιομηχανία εκπέμπει συγκρίσιμες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Παρ' όλα αυτά έχουμε σοβαρά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης αλλά και σε διάφορες περιοχές του κόσμου δεν είναι κάτι που μπορούμε απλά να το αγνοήσουμε. Και νομίζω ότι μια νεκρή θάλασσα δεν είναι σε θέση να επιβιώσει. Γι' αυτό θα πρέπει να εφαρμόσουν την αρχή της προληπτικότητας, διότι οι επιπτώσεις είναι δραματικές όταν περιμένουμε υπερβολικά. Νομίζω ότι η πρόταση είναι αρκετά προσεκτική και ορισμένοι άλλωστε είπαν ότι δεν έχουμε και τόσα πολλά σκάφη υπό ευρωπαϊκή σημαία, επομένως δεν επηρεάζονται και τόσα πολλά, τόσο μεγάλος αριθμός σκαφών. Γνωρίζουμε ότι πολλοί ε, απασχολούν προσωπικό από άλλες χώρες, έχουν σημαίες άλλων χωρών, μπορούμε βέβαια να το συζητήσουμε αυτό. Όσον αφορά ωστόσο τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, να τον ξαναευχαριστήσω θερμά για το γεγονός ότι εξηγήσατε γιατί... Τι ε, δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ε, τα αλλιευτικά ε, σκάφη, αλλά μόνο εκείνα με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 5.000 νομίζω ότι το πεδίο εφαρμογή είναι σχετικά περιορισμένο. νομίζω επίσης ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε μια προθυμία να θεσπιστεί, να θεσπιστούν κανόνες που θα μπορέσουν και να εφαρμοστούν στην πράξη. Το ότι είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο έχει τονιστεί από όλου. Πρέπει να λάβουμε μέτρα. Και αυτό είναι άλλωστε και ο στόχος της πρότασης να δημιουργηθεί μια βάση και να θεσπιστούν φιλόδοξοι στόχοι και στην ναυτιλία. Νομίζω ότι ε, για τις λεπτομέρειες θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και με τους εκπροσώπους των άλλων πολιτικών ομίλων και με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ όλους όσοι πήρατε το λόγο και ε, η ψηφοφορία θα γίνει στην επόμενη μας συνεδρία στις 12 το πεσημέρι και περνάμε τώρα στο ε, τελευταία μας, το τελευταίο μας θέμα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Βαλεάν και το θέμα αφορά τις ηλεκτρονικές συνδιαλέξεις. Ευχαριστώ. Ο κανονισμός αυτός συνοδεύει την απόφαση για την ανάπτυξη του διαλειτουργικού συστήματος e-call σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σας το παρουσίασα στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η γνωμοδότηση εξετάζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Χαιρετίζω αυτή την πρόταση διότι πρόκειται για μια θετική πρόταση και θεωρώ ότι το σύστημα e-call μπορεί να ε, μειώσει σημαντικά τους θανάτους και τους κινδύνους στους δρόμους. Ως εισηγήτρια υποστήριξα την πρόταση για την οποία υπέβαλα κάποιες τροπολογίες διευκρινιστικές σε σημαντικά ζητήματα όσον αφορά για παράδειγμα τους ε, ε, ορισμούς της πλατφόρμας τηλεματικής και αλλού. Όσον αφορά την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού ε, συστήματος. Τα αρχήματα στο μέλλον θα είναι εξοπλισμένο με ε, πλατφόρμες τηλεματικής. Θα διαθέτουν ασύρματη επικοινωνία, τεχνολογία εντοπισμού και τεχνολογία αξιολόγησης. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει και ειδική πρόβλεψη για ευφύ συστήματα όσον αφορά τις πλατφόρμες τηλεματικής. Οι απαιτήσει θα πρέπει να επικεντρώνονται στις λειτουργίες ε, ανάγκη και στην ε, πλατφόρμα 112. Ε, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα νομικό κενό όσον αφορά τις ε, καθυστερήσεις και τη λειτουργικότητα του συστήματος 112. Ζήτησα από την Επιτροπή να προτείνει έναν κατονισμό όσον αφορά τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες πρόσθετης αξίας που μπορούν να ωφελήσουν τους καταναλωτές. Επίσης έχω συμπεριλάβει τροπολογίες που θα δώσουν τη δυνατότητα σε όσους έχουν ήδη κινηθεί να συνεχίσουν να ε, προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ε, καταναλωτές. Επίσης, το e-call σύστημα θα πρέπει να μπορεί να συνεπάρχει με το σύστημα 112 και γι' αυτό έχω ε, συμπεριλάβει ένα σχετικό ε, ορισμό για τα τρίτα μέρη. Ωστόσο, ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να επιλέγει το ένα ή το άλλο το σύστημα. Για την ίση πρόσβαση στην αγορά και στην κάλυψη της αγοράς, τρίτη πάροχη θα πρέπει να επιτρέπεται να ε, επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται εφόσον το σύστημα 112 είναι διαθέσιμο έστω ως δεύτερη επιλογή. Για όλους αυτούς τους λόγους συμπεριέλαβα ορισμούς για το ...η call σύστημα για το δίκτυο, τους δέκτες και τους ε, παραλήπτες. Δεν υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία ως προς αυτά στην αρχική πρόταση, γι' αυτό θεώρησα ότι ήταν σημαντικό. Όσον αφορά την ε, συμβατότητα και τα δορυφορικά συστήματα, νομίζω ότι οι κατασκευαστές δεν θα πρέπει να είναι αναγκασμένοι να συμμορφώνονται με ε, δέκτες, χωρίς να υπάρχει πλήρης διαθεσιμότητα των δορυφόρων εντοπισμού. Έως επιτευχθεί κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική αυτή η απέτηση. Επίσης πιστεύω ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να γνωρίζει όλες τις ε, υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις κατεξοδότητες πράξεις και να έχει τον ενδειγμένο χρόνο για να αξιολογεί τα συστήματά της. Γι' αυτό το λόγο προτείνω ότι η θέση σε ισχύ του συγκεκριμένου κανονισμού θα πρέπει να οριστεί για τον Ιούνιο του 2016. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και για τις προτάσεις τροπολογίας. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Μπέλετ. Uh, Σας ευχαριστώ. Ε. ε, το ΕΛΚ συμφωνεί με τα βασικά στοιχεία της πρότασης γιατί θα είναι πολύ θετική για όλους τους καταναλωτές, για τους οδηγούς, αλλά και, την, και τους συνεπιβάτες. Τώρα, ήδη έχουμε υποβάλει κάποιες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να τις επαναλάβω. Σε ό,τι αφορά τις λύσεις ε, των τρίτων, των τρίτων παρόχων, κατά πόσο είναι κατάλληλη εναλλακτική, η η συγγήτρια έχει καταθέσει την τροπολογία υπαριθμών 7 για διεύρυνση του ορισμού του e για να καλύπτει και άλλα κανάλια. Ε, συμφωνούμε με την προσέγγιση, είναι λογική προσέγγιση. Να έχουμε συνύπαρξη στο μέλλον με το σύστημα e σε αυτό που, το υποχρεωτικό και αυτό που θα στηρίζεται στον αριθμό κλίση 112. Επίσης, έχουμε ένα σύστημα που στηρίζεται στην κινητή τηλεφωνία ενσωματωμένο. Ξέρουμε ότι η, οι τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας μπορεί να είναι πιο προσιτές οικονομικά στον καταναλωτή, αλλά ε, μπορούν ε, να τεθούν εκτός λειτουργίας. Θέλουμε επιπλέον ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί ναι, μεν ε, η κινητή τηλεφωνία μπορεί να γίνει αποδεκτή, αλλά με επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές. Γνωρίζουμε από τους συναδέλφους της ΤΡΑΝ και ΙΜΚΟ ότι οι συγητές απέκλεισαν αυτές τις πιθανότητες, αυτές τις εναλλακτικές λύσεις. Δεν ξέρω αν εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι παρόν για να μας διαφωτίσει για το κατά πόσο ε, είναι εφικτή επιλογή η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας για την περίπτωση του e-call. Ε, σε ό,τι αφορά το θέμα Γαλιλαίο, φυσικά θα πρέπει να είναι προ η σχετική τεχνολογία και συμφωνούμε η εισηγήτρια συμπεριέλαβε τον όρο λειτουργικός, operational, σημαντικό αυτό. Φυσικά θα πρέπει να είναι πλήρη, πλήρως λειτουργικό το σύστημα, αλλά χρειαζόμαστε περαιτέρω προσπάθεια και θα πρέπει να προβλέψουμε μεταβατική περίοδο και να δούμε τι θα συμβεί σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, τι θα ισχύσει. Και τέλος, σημαντικό όμως, είναι το θέμα του Open Access Platform, της πλατφόρμας ε, ελεύθερης ανοιχτής πρόσβασης. Σημαντικό ζήτημα που έχει παραμείνει εκρεμές. Και από τη στιγμή που θα μπει το e-call στα οχήματα και θα σωματωθεί, φυσικά το θέλουμε το συντομότερο δυνατό, θα είναι δυνατό να το αλλάξουμε για να συμπεριλάβουμε τις επιπλέον ε, υπηρεσίες τηλεματικής στο μέλλον. Και επαναλαμβάνω, είμαστε υπέρ μιας ε, ταχεία συμπερίληψη ε, του e αλλά αν επισπεύσουμε τα πράγματα θα είναι δυνατόν να ανοίξουμε μετά αυτό το σχετικά κλειστό σύστημα, ώστε να περιλάβει και άλλες τηλεματικές υπηρεσίες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την αιτιολογική σκέψη 9, όπου αναφέρει ότι θα πρέπει το σύστημα να είναι προσιτό, δωρεάν, χωρίς διάκριση προς όλους τους ανεξάρτητους παρόχους με πλατφόρμες διαλειτουργικές και ανοιχτής πρόσβασης. Πολύ καλά όλα αυτά, αλλά πώς ε, θα το συνδυάσουμε με την άμεση ε, εφαρμογή και μάλιστα ενός σχετικά κλειστού συστήματος. Τι προτείνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και πώς θα υλοποιήσουμε την αιτιολογική σκέψη 9 μέσω και μακροπρόθεσμα. Ίσως θα μπορούσε να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μακροπρό... βράχει πρόθεσμα μάλλον κάποιες ε, επιπλέον τεχνικές προδιαγραφές. Το ζήτημα αυτό επηρεάζει και το χρονοδιάγραμμα γιατί η η συγγήτρια προτείνει εισαγωγή της υποχρεωτικής κλήσης ή call τον Ιούνιο του 2016. Οπότε στο μεταξύ θα μπορούμε να καλύψουμε και το θέμα της ανοιχτής πρόσβασης της πλατφόρμας αυτής. Αυτές λοιπόν είναι οι ερωτήσεις που έχω και προς την εισηγητριά μας και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Πρόντι που εκπροσωπεί τον κύριο Πυρίλο που είναι σκιώδης ηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να διαβάσω ένα έγγραφο που μου παρακάλεσε ο Μάριο Πυρίλο να σας παρουσιάσω σε τούτη τη συνεδρίαση. Η εναρμονισμένη υλοποίηση σε ευρωπαϊκή κλίμακα για μια υπηρεσία e-call, το οποίο να είναι διαλειτουργικό, βρίσκεται στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2005 και αποτελεί μια δράση προτεραιότητας ε, για την ε, δημιουργία συστημάτων ε, ευφυών μεταφορών. Μετά από μια μακρά περίοδο διαβουλεύσεων, η Κομισιόν το περασμένο Ιούνιο υπέβαλε δύο νομοθετικές προτάσεις με στόχο να εισάγει στο σύστημα κοινοτικής τυποποίησης των αυτοκινήτων την υποχρέωση εγκατάστασης εντός το τέλος του 2015 ένα, ένα σύστημα e-call μέσα στο αυτοκίνητο. Στηρίζω και συμμερίζομαι τη θέση της Κομισιόν, την πρόταση της Κομισιόν, εφόσον στόχο έχει να διαχειριστούμε σωστά τα επίγοντα, τα, τις επίγουσες κλήσεις μέσα της εφαρμογής της αρχής του Golden Hour. Για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος θεωρώ ότι είναι απαραίτητο το σύστημα e-call να είναι ενσωματωμένο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, έτσι ώστε η υπηρεσία αυτή να είναι προσιτή και αξιόπιστη και να μην ε, μπορούν να απομακρυνθούν αυτά τα συστήματα, να μην ενεργοποιούνται για για να εγγυηθούμε την πλήρη λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του οχήματο, το σύστημα e-call θα πρέπει να υπόκειται σε λειτουργικά τεστ περιοδικά. Ε, συμμερίζομαι με την εισηγήτρια την ανάγκη ε, η Κομισιόν υποβάλλει μια νομοθετική πρόταση εντός του τέλος του 2014 με στόχο να ρυθμιστεί η βάση για το ε, ηλεκτρονικές κλήσεις. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για μια πλατφόρμα που παρέχει μια δημόσια υπηρεσία επίγουσα, είναι απαραίτητο να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση που να συνοδεύεται από πλήρη προστασία των προσωπικών στοιχείων. Είμαι υπέρ τέλος της δυνατότητας σε σύνδεσης με το e-call πλέον ε, υπηρεσιών, αλλά αυτές οι εφαρμογέ θα πρέπει να εγγυώνται την πλήρη πρόσβαση με στόχο την επισκεφή και συντήρηση της υπηρεσίας ε, πήγους, ε, των επιγόντων μάλλον υπηρεσιών. Εγώ είμαι επιπισμένος, θέλω να προσθέσω, γιατί τον επίγοντα χαρακτήρα αυτής της τεχνολογίας, γιατί προφανώς ο χρόνος που μπορεί να εξοικονομηθεί για μια παρέμβαση στο χώρο του ατυχήματος μπορεί να είναι ε, καθοριστικός. σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα είναι καθοριστικός για να σωθούν ζωές και για να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων που έχουν ε, τραυματιστεί. Το Γαλιλαίο αποτελεί φυσικά μια πρόοδο σε σχέση με το GPS, όμως πιστεύω πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται και τα δύο συστήματα έτσι ώστε να βελτιωθεί και η δυνατότητα και η ακρίβεια του εντοπισμού Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και οι μετρητές επιτάχυνσης που θα πρέπει να δίνονται άμεσα στα τηλεφωνήματα αυτά, ανάλογα με τη σοβαρότητα και το ατυχήματος. Αυτό μπορεί να δίνεται από το ποσοστό μείωση της ταχύτητας αλλά και από τις ε, φυγόκεντρες ε, συνιστώσεις που μπορεί να δώσουν, να δώσουν μια πληροφορία όσον αφορά τι, πόσες βόλτες έχει φέρει το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ατυχήματος. Και αυτές οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στοσενόφσκι. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης ε, εισηγητής ε, της ομάδας συντηρητικών και μεταρρυθμιστών και θα ήθελα εκ μέρους της ομάδας μου να υποστηρίξω την έκθεση καθώς και τις τροπολογίες της εισηγήτριας. Από ό,τι ξέρω, το σύστημα επιγουσών κλήσεων ήδη βρίσκεται ε, σε προχωρημένο στάδιο ώστε να μπορεί να ενσωματώσει και το σύστημα e-call και το επίπεδο τεχνολογικής πρόοδου είναι πολύ υψηλό ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε συμβατότητα με το νέο σύστημα e-call. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Η κυρία Συγήτρια ζήτησε λίγο περισσότερο καιρό για τη φάση της ε, δοκιμής, των δοκιμών του συστήματος και συμφωνώ γιατί θα συμπέσει η εφαρμογή του e-call με την εφαρμογή του συστήματος Γαλιλαίου είναι επίσης περίπλοκο τεχνολογικά θέμα. Γι' αυτό και καλό θα ήταν να αφήσουμε περισσότερο χρόνο για τις δοκιμές. Τώρα έχουμε το ισχύον σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και θα έχουμε και πολλές ε, εναλλακτικέ λύσει στο μέλλον χάρη στι ραγδαίε τεχνολογικέ εξελίξει. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ανοιχτοί, να μην κλείσουμε το σύστημά μα για να μπορούμε να συμπεριλάβουμε στο μέλλον τι νέε τεχνολογίε. Επίση, αν έχουμε λίγο περισσότερο καιρό, θα μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε και τις ε, νομικές πτυχέ τη πρόταση. Γιατί θα πρέπει να δούμε ποιος φέρει την ευθύνη σε περίπτωση που δεν υπάρχει σήμα από τα κινητά. Ποιος θα φταίει, ο πομπός, ο δέκτης, ο πάροχος. Υπάρχουν πολλές νομικές πτυχές του e-call που θα πρέπει να διευκρινιστούν. Και είμαι στη διάθεσή σας για συνεργασία για να καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό σύστημα. γιατί χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο σύστημα για την προστασία των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Οντί έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση έχω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, κάτι που μας επισήμαναν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων. Γιατί πολλά αυτοκίνητα ήδη περιλαμβάνουν αυτόν τον εξοπλισμό στα οχήματά τους. Δεν περίμενα τον κανονισμό για να προτείνω αυτήν την υπηρεσία στους πελάτες τους. Οπότε, από τη στιγμή που οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη στις διαδικασίες α, τις βιομηχανικές αυτή τη δυνατότητα του εξοπλισμού και μάλιστα με καλύτερη ποιότητα από αυτή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσουν να κρατήσουν αυτόν τον εξοπλισμό χωρίς να τροποποιήσουν την βιομηχανική τους διαδικασία για να μην πλήξουμε τους ε, καλούς ε, αυτοκινητοβιομηχάνους που ήδη συμπεριέλαβαν στα οχήματά τους τέτοιο, τέτοια δυνατότητα. Ο κύριος Οντερστάλερ είναι ο εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε, ε, σας έχουν υποβληθεί πολλές ερωτήσεις και από τον κύριο Μπέλετ, τον Ντί και άλλους. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να Ευχαριστήσω την Επιτροπή ΤΡΟΕΜ για την γνωμοδότησή της όσον αφορά τη γνωμοδότησή της για το σύστημα e-call. Χαιρετίζουμε και τη θέση του εισηγητή ότι ο κανονισμός e-call θα πρέπει να εστιάζεται στις ε, ε, επίγουσες υπηρεσίες στο πλαίσιο των υποδομών 112 για να μην δημιουργηθούν νομικά κενά όσον αφορά τις ευθύνες. Η συμπερίληψη μιας πλατφόρμας τηλεματικής στην λίστα προτεραιοτήτων της ε, οδηγίας ITS, ωστόσο θα ε, απαιτούσε αναθεώρηση της οδηγίας αυτής. Επομένως η προθεσμία για το 2014 θα ήταν ανέφικτη. Επίσης δεν είναι σίγουρο αν θα πρέπει να, ότι θα μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένες προδιαγραφές για ένα τέτοιο σύστημα. Όσον αφορά τους ορισμούς, η Κομισιόν χαιρετίζει την προσπάθεια να ε, αποσαφινιστεί το κείμενο, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την απόκληση από ε, υφιστάμενους ορισμούς όπως, ο 300, όπως αυτός που περιλαμβάνεται στο 305 κάτω του 2013. Για το Γαλιλαίο και το Έγνος. Οι υπηρεσίε αυτές θα είναι διαθέσιμες ήδη από το 2013, 2014 με συγχωρείτε, και θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της συμβατότητας των συστημάτων αυτών. Επίσης, ε, πομπή και δέκτες με πολλά τσίπ ε, γίνονται όλο και πιο συνήθις. Η Κομισιόν έχει κάποιες ανησυχίες για τις τροπολογίες 5 και 18 αφού το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι μη ιχνηλάσιμο αν θέλουμε να ε, σεβόμαστε τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά τι κινητές συσκευέ, η πρόταση δεν αποκλείει τη χρήση κινητών συσκευών, αλλά θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και αυτό θέτει ορισμένα ερωτήματα στο πλαίσιο της χρήσης των κινητών συσκευών. Πρώτον θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ε, μια τέτοια συσκευή θα είναι παρούσα στο όχημα, ότι θα είναι ανθεκτική σε προσκρούσεις σε περίπτωση τροχαίου και επίση θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτέ οι κινητέ ε, συσκευέ θα είναι λειτουργικέ, θα είναι φορτισμένε και επίση θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τεχνικέ υπηρεσίε θα μπορούν να ελέγχουν τέτοιου είδου συσκευέ, αφού δεν είναι καθεαυτές τμήμα του οχήματο. Για το ερώτημα για τα υπάρχοντα συστήματα, αυτά που ήδη δηλαδή σε πολλού κατασκευαστέ συμπεριλαμβάνονται στα οχήματα που παράγονται, η απέτηση για το 112 το e-call αφορά νέους τύπους, νέα μοντέλα. Άρα δεν αφορά τα οχήματα που έχουν ήδη κατασκευαστεί και φυσικά μπορούν οι κατασκευαστές από εδώ και πέρα κατά το σχεδιασμό νέων οχημάτων να λάβουν υπόψη τους ε, τις απαιτήσει όσον αφορά το σύστημα 112 e-call. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τώρα να δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Βαλεάν, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους και την γενική υποστήριξη της έκθεσης και των τροπολογιών. Νομίζω ότι καλύψαμε τα πιο ουσιώδη σημεία και σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι ποιο είναι το νευραλγικό σημείο του κανονισμού. Σε ό,τι αφορά τις ε, τεχνολογίες, ε, να συμφωνήσω, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε αν γίνεται πραγματικός εντοπισμός της θέσης με τα κινητά. Γιατί Ζητήσαμε, απαιτείται ήδη από τα smartphones να μπορούν να δίνουν τον εντοπισμό της θέσης όταν γίνεται κλίση με βάση τον αριθμό κλίση 112. Οπότε θα ήταν τέλειο να έχουμε μια εναρμονισμένη προσέγγιση και να ισχύει και για τα smartphones και για τα ε, και στα αυτοκίνητα με, την, ε, με τις συσκευές. Σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα ανοιχτή ε, πρόσβασης, είμαι σίγουρη ότι αυτή η πλατφόρμα είναι το μέλλον. Και θα είναι και ένα σημαντικό επιχειρησιακό μοντέλο για την καλύτερη συνδεσιμότητα. Και με τις νέες τεχνολογίες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα έχουμε ωφέλη για όλους. Οπότε αυτό είναι το μέλλον και θα πρέπει να το υποστήριξουμε. Απ' την άλλη, όπως είπα εγώ και επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε θέματα ευθύνης, προστασίας των δεδομένων. Οπότε, αν στον κανονισμό αυτό συμπεριλάβουμε και την πλατφόρμα ανοιχτή πρόσβασης, θα δημιουργήσει ε, επιπλοκές και ίσως και καθυστερήσεις. Ενώ στην ουσία μιλούμε για μια πλατφόρμα για επίγουσες κλήσεις. Πάντως πιστεύω ότι οι σχεδιαστές και κατασκευαστές αυτοκινήτων καθώς και οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ήδη έχουν υπόψη τους ότι αυτή η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες υπηρεσίες. Οπότε θα έρθει φυσιολογικά, θα έρθει από μόνη της. Ήδη προλυαίνεται το έδαφος για αυτή την πλατφόρμα. Τώρα θα είναι ανοιχτή ή όχι και ανοιχτή γιατί και για ποιον και ποιος είναι υπεύθυνο ποιος θα είναι ο ελεγκτής ε, και ποιος θα διαχειρίζεται τα δεδομένα, ποιος θα τα επεξεργάζεται, όλα αυτά νομίζω ότι καλύτερα αποτελέσουν το αντικείμενο άλλου κανονισμού. Αν το θεωρεί πρόημο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 20 Απριλίου του 2014, μπορεί να μην έχει και άδικο. Το θέμα είναι όμως ότι η αυτοκινητοβιομηχανία μας ε, ζητά αυτό το χρονοδιάγραμμα. Πολλοί ενδιαφέρονται από πολλούς και διάφορους κλάδους για τις διευκρινήσεις για το πώς θα λειτουργεί αυτή η ανοιχτή πλατφόρμα για να μπορέσουν να προετοιμάσουν τα νέα τους ε, επιχειρηματικά μοντέλα. Επαναλαμβάνω ευχαριστώ θερμά τους ε, συναδέλφους για τα σχόλιά τους και προσβλέπω σε συνέχιση τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Βαλέαν και ευχαριστώ φυσικά και τους υπόλοιπους συναδέλφους ε, Προθεσμία για τις τροπολογίες. Λίγη στις 5 Δεκεμβρίου το μεσημέρι. Ουσιαστικά δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης που προβλέπει την ενημέρωση για δύο τριμερείς διαλόγους ε, που αφορούν σημαντικά θέματα. Ε, το πρώτο αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών έκθεση το Σενόφσκι, το ψηφίσαμε και υπάρχει διαπραγματευτική εντολή με βάση της, την πρωινή ψηφοφορία. Κύριε Σενόφσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όντως, ψηφίσαμε σήμερα για το ευρυζωνικό διαδίκτυο σήμερα το πρωί και ο τριμερής διάλογος που έγινε και μετά τη σημερινή ψηφοφορία ολοκληρώνεται μία μακρά περίοδο με, τη σημερινή ψηφοφορία ολοκληρώνεται μία μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων που κράτησε σχεδόν μία διετία. Έγινε ο τριμερής διάλογος, ήταν ε, απαιτητικός και στην τελευταία συνεδρία του τριμερούς διαλόγου ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις Ξεκινήσαμε 7 το πρωί και τελειώσαμε σχεδόν τα μεσάνυχτα. Ήταν αρκετά επαχθής ε, διαδικασία και δυσχερής ε, η διαπραγμάτευση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την κυρία Άντερς, τότε τον κύριο Κρότσμαν και πολλούς άλλους που συνέβαλαν στην διαδικασία και χάρη στην άοκρη προσπάθεια των κυρία, της κυρία Στράουτμαν και του κυρίου Χάκμαν που ακούραστη εργάστηκαν για ένα πεντάωρο συναπτό, καταφέραμε να καταλήξουμε στη συμφωνία. Και τελικά το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου έγινε δεκτό από το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ θερμά για την αγαστή συνεργασία που είχαμε με όλους τους συναδέλφους στην Επιτροπή αλλά και με την νομική υπηρεσία, με το, τους υπαλλήλους μας, συνεργάτες μας γιατί υπήρχαν κάποια δύσκολα νομικά ζητήματα. Γιατί εδώ μιλούμε για μια επταετή διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει τα ρυθμίσαμε όλα αυτά και σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας. Γιατί επιτέλους διεκπαιρεώσαμε αυτό το θέμα, μπορούμε να το παραπέμψουμε στην Ολομέλεια. Δεν ξέρω αν θα είναι η Ολομέλεια του Ιανουαρίου ή του Φεβρουαρίου, Πάντως το ζήτημα είναι έτοιμο για την Ολομέλεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την Λιθουανική Προεδρία για τις προσπάθειές τους, γιατί πραγματικά ήταν ανεκτήμητη η συμβολή τους και χάρη στη δική τους συνεργασία μπορέσαμε να ρυθμίσουμε κάποια ζητήματα που αρχικά ήταν λίγο αόριστα. Επαναλαμβάνω, το ο τριμερής διάλογος διεκπαιρεώθηκε και με τη σημερινή ψηφοφορία ολοκληρώσαμε και το δικό μας έργο Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους που ξόδεψαν ώρες ολόκληρες στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ε, και φυσικά ολόκληρη Επιτροπή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά εσάς κυρία Τωσενόφσκη που συμβάλλετε και εσείς ως συγκεκριτή στη διεκπαιρέωση αυτού του θέματος. Η κυρία Ολσκοκ για ένα άλλο σημαντικό θέμα. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να σας πω για το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε τον πρώτο τριμερό ε, διάλογο για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση στις 27 Νοεμβρίου, αυτή τη βδομάδα δηλαδή. Και η Λιθουανική Προεδρία βεβαίως παρέστη. Και σε, αυτή την πρώτη, σε αυτό τον πρώτο τριμερό, τριμερή διάλογο επί Κεντρωθήκαμε στα άρθρα 1 και 9 που αφορούν την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και στα άρθρα 1 έως 19 ε, που αφορούν τις ε, trust services τις λεγόμενες. Το θέμα αυτό μας ακολουθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα προγράμματα και πυρήνας του είναι να προσπαθήσουμε να ενιοποιήσουμε τα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα κράτη-μέλη. Διότι κάθε κράτος μέλος έχει αναπτύξει ένα δικό του σύστημα και αυτά τα συστήματα όλα σκοπός είναι να ενιοποιηθούν διότι δεν είναι διαλειτουργικά. Θέλαμε να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να φροντίσουμε ώστε οι συναλλαγές μέσω ίντερνετ να γίνουν πιο ασφαλείς. Μπορεί για παράδειγμα να γίνει μια ανταλλαγή μεταξύ διαφορών ευρωπαϊκών ε, αρχών ή υπηρεσιών. Τα πάντα στην ουσία μπορεί να αφορά κάτι τέτοιο αλλαγή διεύθυνσης ή αίτηση για ε, θέση σε πανεπιστήμιο, αλλά σκοπός επίσης είναι να προωθηθεί και το εμπόριο. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει κάποιο σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που θα επιτρέπει την αλληλοκατανόηση και ταυτόχρονα θα διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Αυτό είναι, με λίγα λόγια, το υπόβαθρο για αυτήν την εξέλιξη στον ε, τεχνολογικό κόσμο που ζούμε σήμερα. Ε, ο επόμενο τριμερή διάλογο θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου και νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούμε άλλη μία ημερομηνία διότι τα ζητήματα αυτά βεβαίως είναι πολύ περίπλοκα για το Συμβούλιο και το Συμβούλιο δεν είναι απαραίτητος ε, της ίδιας γνώμης με εμάς. Έχουμε, ωστόσο πιστεύω ότι θα βρούμε μια λύση. Έχουμε πολύ στενή προθεσμία. Αν θέλουμε στην παρούσα θητεία να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα θα πρέπει έως το, τα μέσα Φεβρουαρίου να το κάνουμε για να το στείλουμε στην Ολομέλεια τον ε, Απρίλιο. Η Λιθουανική Προεδρία σε κάθε περίπτωση ήταν πάρα πολύ Ενεργεί το ίδιο και η Κομισιόν. Και είπαμε και στο, στον προηγούμενο τριμερή διάλογο ότι και η ελληνική προεδρία θα πρέπει επίσης να μας βοηθήσει ώστε να όταν θα αναλάβει τη σκητάλη στις αρχές του επόμενου χρόνου διότι ο τριμερός, τριμερής αυτός διάλογος θα συνεχιστεί και μετά τη Λιθουανική Προεδρία και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα θα βγουν ομαλώς. Είναι πολύ σημαντικό το νομοθέτημα αυτό. Ελπίζω πραγματικά να το καταφέρουμε εντός αυτής της θητείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ολσκοκ είμαστε στο πλευρό σας και εμείς θέλουμε να διεκπαιρεωθεί το θέμα αυτό στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία. Και νομίζω ότι έχουμε μεγάλες πιθανότητες να τα καταφέρουμε. Ολοκληρώνεται η συνεδρίαση. Μην ξεχνάτε ότι στις 3 έχουμε μια πολύ σημαντική ακρόαση για τις τηλεπικοινωνίες και την εσωτερική αγορά των τηλεπικοινωνιών. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και ραντεβού στις 3.